Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την συνεδρίασή μας. Και περνάμε στο σημείο 8 περιμένουμε όμως ένα λεπτό. Το 8. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Πρόκειται για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις υποεξέλιξη, τους υποεξέλιξη τριμερούς διαλόγου, τριμερείς διαλόγους. Και μέχρι σήμερα είχαμε έναν, την, την έναρξη τριμερούς διαλόγου για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Έγινε χθε αυτός ο τριμερής διάλογος. Θα θυμόσαστε, τρεις τομείς είχαμε, στους οποίους ε, τροπολογίες είχαμε εγκρίνει. Τεχνικού χαρακτήρα πρώτον, προσαρμογή της νομοθεσίας ε, με την ε, με τα χρόνια που πέρασαν. Δεύτερον, αν κατεκτέλεση νομικές πράξεις ή κατεντολή νομικές πράξεις πρέπει να ακολουθήσουν. Αποφασιστικό αίτημα από πλευράς μας και πολιτικό ερώτημα, πολιτικός προβληματισμός στην ημερήσια διάταξη. Πώς αυτή η διαδικασία στα Δυτικά Βαλκάνια θα διαμορφωθεί και πώς θα ενταχθεί. Για τα διάφορα θέματα ανταλλάξαμε απόψεις. Ήταν κάπως απογοητευτική η κατάσταση επειδή δεν είχε αυθεντική εντολή διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Ήταν μόνο σε θέση κάποιες τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες να δεχτεί ή να συζητήσει. Και ουσιαστικά μία από τις ε, εννέα όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα της κατεξουσιοδότηση πράξης δεν υπήρξε καμία κίνηση, κινητοποίηση από το Συμβούλιο και το είπα ξεκάθαρα στο Συμβούλιο ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό από εμά ως κατάσταση και έχουμε μια πιθανότητα να προχωρήσουμε μόνο όταν θα έχει το Συμβούλιο εντολή διαπραγμάτευσης και με αυτό το μήνυμα πέρασα να το διαβιβάσουν στο Συμβούλιο και στις 22 Σεπτεμβρίου θα τα ξαναπούμε και θα δώσουμε συνέχεια στον τριμερή διάλογο. Επ' αυτού έχετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες παρεμβάσεις. Δεν έχετε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι το 9. Η γνωμοδότηση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής για την έκθεση για την Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση που έγινε και τώρα έχουμε το σχέδιο του εισηγητή που είναι στα χέρια μας. Έχει τον λόγο εισηγητής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού. Λογικό είναι ότι περιορίστηκα σε ένα μικρό εύρος θεμάτων και αντίστοιχα από δική μας πλευράς θα κατατεθούν τροπολογίες βέβαια ώστε να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί αυτό το πλαίσιο. Στο σχέδιό μου προσπάθησα μια κάποια συνένεση να επιτύχω μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Σίγουρα δεν είναι μια καθαρή γνωμοδότηση της δικής μας ομάδας μόνο. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ σε περαιτέρω βήματα θα βρούμε κοινούς συμβιβασμούς, συμβαστικές λύσεις οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, η ενεργειακή ασφάλεια στην τροφοδότηση, η ανταγωνιστικότητα και η αηφορία πρέπει να είναι αυτοί οι στόχοι. Αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους υλοποιήσουμε να μειώσουμε τις ανάγκες μας ενεργειακά και από την άλλη πλευρά να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες αηφόρες πηγές ενέργειας θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε ώστε από κοινού με συμβάσεις ενεργειακές με τρίτες χώρες από κοινού να διαπραγματευτούμε. Από κοινού είναι σημαντικός ο όρος αυτός. Η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι σημαντικός στόχος και έχει μεγάλη εμβέλεια. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Κοινές προδιαγραφές και τεχνολογίες να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα με την Κίνα εδώ βλέπουμε την τεχνολογία της αποθήκευσης ενέργειας ως ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για να περάσουμε σε ένα περιβάλλον που θα έχει μικρότερη επιβάρυνση από τον άνθρακα. Και αυτά τα σημεία δεν έχουν τόσο έντονα τονιστεί μέχρι τώρα, αλλά στις ανανεώσιμες ενέργειες θέλουμε να περάσουμε στο πάνω από 30% η αποθήκευση ε, της ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας, αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα. Τα τεχνικά συστήματα έχουν εκπονηθεί, τεχνολογικά έχουν δοκιμαστεί, τώρα θα πρέπει τα προσκόμματα και τα εμπόδια να αρθούν για να προχωρήσουμε. Επενδύσεις σε μέτρα αποδοτικότητας ενέργειας, μέσω της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σχέση για παράδειγμα με τους εταίρους μας πρέπει να αυξηθεί η αποδοτικότητά μας. Η θέση μας στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας και στα ανανεώσιμα πρέπει να προχωρήσει, να επεκταθεί. Να σκεφτούμε τι γίνεται με το εξωτερικό εμπόριο και στις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων και τιμών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο. Η πολιτική συνέπεια και συνεκτικότητα στο εξωτερικό εμπόριο έχει μεγάλη σημασία στον ενεργειακό τομέα. Θα ήταν υποκριτικό αν εσωτερικά απαιτούσαμε υψηλές προδιαγραφές, όμως στο εξωτερικό εμπόριο δεν τηρούσαμε αυτές τις προδιαγραφές εμείς οι ίδιοι. Στην Ευρώπη εκφραστήκαμε δεσμευτικά για την μείωση των εκπομπών ρήπων του θερμοκηπίου και δεν είναι δυνατόν η ευθύνη μας, την ευθύνη μας να την απεμπολίσουμε έχοντας ρηπαίνουσα ενέργεια που θα ε, επιβαρύνει το περιβάλλον. Τώρα θέλω να ακούσω ποια είναι τα στοιχεία που σχεδιάζουν να προωθήσουν οι συνάδελφοι και να τα εντάξουμε στο σχέδιο αυτό. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα έχουμε. Ευχαριστώ. Σκιώδεις εισηγητές ακολουθούν. Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, Eh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως ο συνάδελφος ε, Σαλβατόρε Τσίκο δεν μπορεί να παραστεί, μου ζήτησε να παρέμβω και θα το ε, κάνω εγώ. Ζητεί στα Ιταλικά. Τα κλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλέ. Γι' αυτό καλούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενωσιακά να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουμε ασφαλή βιώσιμη ενέργεια και σε χαμηλές τιμές. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 90% του ε, αργού πετρελαίου και το 66% του φυσικού αερίου. Το 94% των μεταφορών εξαρτώνται από πετρελαιοειδή, τα οποία εισάγονται κατά 90%. Μέσω μιας ε, συγκριτικής ανάλυσης προκύπτει επιπλέον ότι στην Ευρώπη οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου είναι υψηλότερες κατά 30 και 100% σε σχέση με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αναλυθεί φιλόδοξη ευρωπαϊκή δράση που θα επιτρέψει να παρέχονται στους καταναλωτές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οικογένειες και επιχειρήσεις ασφαλής ενέργεια, βιώσιμη και ανταγωνιστική. Για αυτό το σκοπό πρέπει να υλοποιήσουμε σημαντικούς μετασχηματισμούς του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος που θα επιτρέψουν στις ροές ενέργειας να διέρχονται ελεύθερα από τα σύνορα, ειδικότερα στα σημεία που αποτελούν σημαντικούς διαδρόμους ε, ενεργειακών δικτύων. Μια φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να επιτρέψει στους καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά. Είναι σημαντικό να αφήσουμε πίσω μας το σημερινό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από το συντονισμό πολλών εθνικών πολιτικών, από φραγμούς αγοράς και από ενεργειακές νησίδες. Επίσης είναι σημαντικό να υλοποιήσουμε το στόχο του 2020 για το 10% βελτιώνοντας ε, την κατάσταση σε 12 κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή διασυνδέονται κατά λιγότερο από 10% όπως Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Κύπρος και Μάλτα. Μεταξύ αυτών πρέπει να συνδεθούν και οι απομονωμένες νησιωτικές περιοχές που χρειάζονται άμεσα την ανάληψη δράσεων στον τομέα των υποδομών με στόχο την προμήθεια ενέργειας. Μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική θα βασιστεί σε χρηματοδοτικά μέσα για την πραγματοποίηση των ε, προγραμμάτων διασύνδεσης όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014. Για να ολοκληρώσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκοπό να βελτιώσει την ικανότητά της ε, να αναδειχθεί στις παγκόσμιες αγοράς ενέργειας μέσω μιας ισχυρής ε, πολιτικής εμπορικής χωρίς αποκλεισμούς. Γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να συνάψουμε εμπορικές συμφωνίες ε, με ρήτρε προνομιακής πρόσβασης στους πόρους μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγών και επενδύσεων δυναμικού με τις χώρες και τις περιοχές που αποτελούν σημεία, στρατηγικά σημεία προμηθειών όπως η Αλγερία, η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μέση και η Αφρική. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Για τους σοσιαλδημοκράτες είμαι εγώ ίδιος ο, εισηγη... ο σκιώδης εισηγητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Σημαντικά στοιχεία εμπεριέχονται στο σχέδιο ψηφίσματος. Εγώ θα ήθελα τρεις συμπληρώσεις να γίνουν. Ο πρώτος τομέας είναι το θέμα των ενεργειακών συμφωνιών. Ο κύριος Φίσας το ανέφερε πιο πριν. Πρέπει ακριβώς ε, στην ευθύνη μας ως ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να καταστήσουμε σαφές ότι οι, τα τμήματα αυτά μιας ενεργειακής εμπορικής συμφωνίας, δηλαδή ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στις εμπορικές συμφωνίες για την ενέργεια πρέπει να συμπεριληφθεί, πράγμα το οποίο αναφέρει ότι οι στόχοι μας για τον ανεφοδιασμό αλλά και οι προδιαγραφές ποιότητας πρέπει να θεσπιστούν και θέλουμε να προαγάγουμε το θέμα των ανανεώσιμων ενεργειών, πηγών ενέργειο, ενέργειας και την αποδοτικότητα της ενέργειας να την βελτιώσουμε επίσης ώστε μέσω της συνέργειας μέσω των κεφαλαίων αυτών για την ενέργεια σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες να έχουμε ένα βαθμό υποστήριξης για την ενεργειακή πολιτική μας. Δηλαδή κάπως πιο διεξοδικά να τονίσουμε τη σπουδαιότητα των θεμάτων της ενέργειας ε, στα αντίστοιχα κεφάλαια μια τέτοια συμφωνίας. Και αυτό με τροπολογίες πρόκειται να το καλύψω ώστε να προχωρήσει. Μετά το σημείο 7, το σημείο της ε, συνεργασίας θα ήθελα με μεγαλύτερη σαφήνεια να αναπτυχθεί αυτό. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι ενεργειακές συμβάσεις και συνθήκες που έχουμε πρέπει να επανεξεταστούν. Έχουμε διμερείς τέτοιες συμφωνίες ως κράτη-μέλη με διάφορες χώρες. Και αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό συμφέρον της Ευρώπης συνολικά, έχω αμφιβολίες γι' αυτό και πρέπει να δούμε την συνολική κατάσταση όταν έχουμε τέτοιες συμβάσεις. Και κατά τούτο πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει για το μέλλον της ολοκλήρωσης, της σύναψης τέτοιων ενεργειακών συμφωνιών. Έχουμε και νομοθεσία που πριν από την κρίση της Ουκρανίας ε, είχε ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και σε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν πολύ επιφυλακτικά και διστακτικά τα κράτη-μέλη όσον αφορούσε την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύναψη τέτοιων συμβάσεων. Τώρα με τα γεγονότα και τα όσα συνέβησαν άλλαξε η κατάσταση και ο Πολωνός Πρωθυπουργό το ζήτησε αυτό. Αυτές οι συμφωνίες, οι συμβάσεις να συνάπτονται κοινοτικά ώστε να έχουν κοινοτικό χαρακτήρα και έτσι πρέπει το θέμα <clears throat> της αναθεώρησης της ενισχύ νομοθεσίας για τέτοιες συμβάσεις να εξεταστεί, να δούμε τι θα γίνει και μια προθεσμία για μια τέτοια αναθεώρηση προβλέπεται, αλλά και κριτήρια για την σύναψη μελλοντικών ενεργειακών συμφωνιών που πρέπει να υπάρξουν και να λειτουργήσουν ώστε να έχουμε μια συνεκτικότητα, ένα συνεκτικό πλαίσιο και οι δράσεις μας ε, να είναι συνεπέστερες. Και έτσι λοιπόν στο 7 ένα νέο σημείο θα προσθεθεί για να δούμε ποια στοιχεία θα αποτελούν μια τέτοια σύμβαση για την ενέργεια από πλευράς μας μελλοντικά. Και η αμοιβαιότητα και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Να υπάρχει δηλαδή ανταπόκριση και αντιστοιχεία μεταξύ των δράσεων των εταίρων. Αμοιβαιότητα και για τις προδιαγραφές αλλά και για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα τρία μου σημεία και τώρα εσείς. Παρακαλώ. Thank Μιλώ εκ μέρους του, του κυρίου Κομόρ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανε ο Πολλά δέχεται η ECR. Το να έχουμε πιο αποτελεσματική αγορά, ε, αυτάρκη αγορά, ε, καλύτερη σχέση κόστους-οφελίας για να βελτιώσουμε την πρόσβαση επίσης, ε, στην πρόσβαση ε, και στις αγορές είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ο ανεφοδιασμός της ενέργειας και να μειώσουμε την εξάρτηση από τα επιμέρους σημεία ανεφοδιασμού. Η πρόθεση του ρόλου του εμπορίου και οι σημαντικές μελλοντικές τεχνολογίες είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία θα θέλαμε να συμπεριληφθούν. Πρώτον, η σημασία της εχώριας ε, ενεργειακής ε, παραγωγής και πόρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το ρόλο του ΠΟΕ και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει παγκόσμια διακυβέρνηση, διεθνείς συμφωνίες και υποστήριξη. Θα έχει μεγαλύτερη νομική σταθερότητα κάτι τέτοιο και θα αυξήσει θα μειώσει συγγνώμη, τις διεθνείς εντάσεις. Ο ΠΟΕ είναι το καταλληλότερο φόρουμ για να συζητηθούν αυτά τα πράγματα και θα ήθελα αυτό να το αντικατοπτρίζει η ΕΝ, η γνωμοδότηση. Επίσης, ε, υπάρχουν τα 13 μέλη του ΠΟΕ ε, που μπορούν να συμφωνήσουν για τα ενεργειακά προϊόντα και τις τεχνολογίες. Ε, θα μπορούσαν έτσι να προστατεύσουμε το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα Υποτίθεται ότι οι συζητήσεις θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος ε, του 2015. Ο επόμενος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω δύο-τρία σημεία. Καταρχά, να πω στον εισηγητή ότι συμφωνώ απόλυτα. Είμαι στο ίδιο μήκο Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε την εξάρτηση από τι εισαγωγέ. Όχι μόνο γιατί ε, εισάγουμε βρώμικη ενέργεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κλίμα, αλλά για να είμαστε αυτόνομοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να είναι ανεξάρτητη η Ευρώπη και γιατί είναι στρατηγική σημασία κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στην έκθεση. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, όπως υπάρχουν ζώνες συγκρούσεων και αποσταθεροποίησης, το θέμα της ε, ενεργειακής αυτονομίας το θέμα της ε, ενεργειακής ανεξαρτησίας θα είναι πολύ σημαντικό τα επερχόμενα χρόνια. Επίσης, σύμφωνο με όλα όσα είπε ο συγητής, θα πρέπει να έχουμε παραγωγή καθαρών ενεργειών, οικονομία, οικονομία ενέργειας, ε, καινοτομία, καλύτερο συντονισμό των εθνικών μας πολιτικών. Όλα αυτά καλά είναι. Αλλά εγώ τονίζω το εξή σημείο. Είναι στρατηγική σημασία η Ευρώπη να αποφασίσει να έχει το συντομότερο δυνατόν μια πλήρη και απόλυτη ενεργειακή αυτονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για ένα καλό έγγραφο εργασίας και για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας είναι σημαντική υπόθεση είναι η δεύτερη αυτή προσέγγιση και για τα, τα προτινόμενα στο σχέδιο και στις διατυπώσεις ε, συμφωνώ και το σχέδιο αυτό είναι ισορροπημένο. Τώρα, αν εγώ θα είμαι εκείνο ο οποίος θα τα πει ότι όλα είναι σωστά, έχω και κάποιες ε, επιφυλάξεις. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για το σημείο 2, για το ενεργειακό κεφάλαιο, που είμαι υπέρ να έχουμε ένα ενεργειακό κεφάλαιο σε συμβάσεις ε, εμπορίου, αλλά είμαστε κατά της ε, εισαγωγής fracking gas ή όσον αφορά από τα πισούχα, ασφαλτούχα κοιτάσματα θα πρέπει να εκφράσουμε πώς θα, έχουμε, διαμορφώσουμε τη συνεργασία μας σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προσέγγισή μας. Διότι αν καθυστερήσουμε και παραμείνουμε στις προσεγγίσεις των μεγάλων ε, ενεργειακών επιχειρήσεων, ε, τότε δεν θα είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί. Να μην εκπλησώμεθα ότι οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις λοιπόν δεν θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η ευφυής ε, φορολόγηση των προϊόντων αυτών θα έχει πραγματικά ε, μέλλον και γι' αυτό στη γνωμοδότησή μας όσον αφορά και την Επιτροπή Βιομηχανίας στην ε, διατύπωση των πολιτικών για την, τα ενεργειακά αυτά προϊόντα από πλευράς της έρευνας και της ανάπτυξης πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και να προσεγγίσουμε έτσι αυτά τα θέματα για να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια και συνεκτικότητα με τις άλλες πολιτικές μας. Υποστηρίζω τη θέση του ε, εισηγητού για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και να έχουμε μια πιο διαφανή παρουσίαση των, του κόστους ε, στην Γερμανία έχουμε, γνωρίζουμε πόσο ακριβή είναι η εκμετάλλευση των πυρηνικών αντιδραστήρων και εδώ επιβαρύνονται και μελλοντικές γενναίες σε σχέση με την ε, ε, ε, επιβάρυνση αυτή και ιδιαίτερα όσον αφορά την ισορροπημένη προσέγγιση από πλευράς μας όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια ελπίζω ότι θα μπορέσουν να κατατεθούν περαιτέρω τροπολογίες ώστε να συμπληρώσουμε κάποια θέματα θα υποστηρίζαμε ένα τέτοιο εγχείρημα όμως ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αν είμαστε να μην ακολουθήσουμε μια μη ελεγχόμενη ε, πορεία σε σχέση με το, την κερδοφορία και το, την επιβάρυνση κόστους βλέπουμε ότι και από πλευράς των Ρώσων και των ΙΠΑ και του αραβικού κόσμου υπάρχει αυτό το στοιχείο. Και για ένα κονσόρτσιο Πολωνών, Βρετανών ε, και άλλων όσον αφορά την περιοχή του Σαβιάνσκ με την επισήμανση ότι για την παραγωγή αερίου μέσω διαρρογμάτωσης, ε, υδραυλικής ε, διαρρογμάτωσης, ε, γνωρίζουμε για ποια πράγματα γίνεται λόγος εδώ και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε συμφέρον όσον αφορά την εκμετάλλευση, την μείωση της εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων. Πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, ακόμα και σε χώρες όπως η Ελλάδα που η υποστήριξη της, ε, ηλιακής, ε, της εκμετάλλευσης ε, της ηλιακής ενέργειας θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και σε σχέση με την Επιτροπή Ενέργειας να λάβουν υπόψη περισσότερο τις δικές μας απόψεις ώστε να αποφύγουμε αποτυχία στην Ολομέλεια μιας νέας έκθεσης που θα τεθεί εκεί σε ψηφοφορία προς έγκριση. Ευχαριστούμε και συμμεριζόμαστε αυτή την ελπίδα. Ο κύριος Μπορέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ενεργειακό θέμα θέτει την Ευρώπη έναντι δύο προκλήσεων. Η πρώτη εσωτερική και αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την εσωτερική αγορά, που είναι κατακαιρματισμένη. Το δεύτερο αφορά την, το εξωτερικό θέμα, την εξωτερική διάσταση και την εξωτερική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το κείμενο αυτό μιλάει πολύ για το θέμα του κόστους, ε, το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και την πρόθεση ενεργειακών διέργειας. Ε, συμφωνούμε από αυτόν. Θέλουμε όμως παράλληλα να θέσουμε την ε, προσοχή σας ε, πάνω στο εξής. Οι ενεργειακές υποδομές και ανανεώσιμες τι σημασία έχουν για την Ευρώπη και για τις τοπικές κοινότητες. Η αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να δώσει, να είναι η αφορμή για τοπικέ πολιτικέ ενέργειε. Όταν μιλάμε για θεκτικότητα και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά το κόστο, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη και αυτό ε, πώ ξεκινάει από σωστή εκπαίδευση των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων. Και μη βιώσιμοι τρόποι ζωή αυξάνουν το κόστο, αλλά και πλήττουν α, τον πλανήτη. Η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει ε, ένα ρόλο μεταξύ προβληματικών γεωπολιτικών ισορροπιών ε, δεν θα πρέπει να αισθανθούμε πιο ευάλωτοι. Ε, πέρα από την Νορβηγία, την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν, υπάρχουν και νέες γεωγραφικές περιοχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της, όπως ε, στην Κεντρική Ασία, κυρίως το Καζακστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει αυτές τις στρατηγικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες συνθήκες και την κρίση με την Ρωσία, τον σχέση με τη Ρωσία. Πολλά από αυτά τα θέματα θα παραμείνουν στην ατζέντα της Επιτροπής μας και στο εγγύς μέλλον. Θα επιμείνω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα της ε, γνωμοδότησης που σήμερα συζητάμε. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα που αναφέρθηκε στο αρχικό σημείο της, ε, του κειμένου της Κομισιόν θεωρείται ως ε, εξετάσει από τη σκοπιά των ενεργειακών πηγών. Μην ξεχνάμε όμως και το ρόλο που έχουν οι πολίτες μας εδώ. Η ευαισθησία αυτή ε, συνδέεται και με αυτό που λέει το σημείο 4, δηλαδή το, ο περιορισμός της ενεργειακής ζήτησης. Στο τρίτο σημείο, αφορά, το τρίτο σημείο αφορά την ενεργειακή πολιτική μας και είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Και αυτό ε, μας αναγκάζει σε ένα προβληματισμό για τις νέες αγορές. Ε, κατά τη διάρκεια της θητείας μας ε, θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τις αναδυόμενες αγορές, ε, λαμβάνοντας υπόψη την, παρακολούθηση του Monitoring Group ε, των χωρών της Κεντρικής Ασίας. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης το ρόλο που, θα έχει, που έχει και θα έχει η Ρωσία και η Ουκρανία. Στο σημείο 5, μία σύντομη αναφορά σε έμεσους, τους έμεσους παράγοντες που αναφέρει ο εισηγητής. Το, έχουμε το, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πέρα από αυτά πρέπει να δούμε τι επίπτωση έχουν και οι δομές, οι υποδομές στην, στο έδαφό μας. Εδώ μιλάμε για χρήσιμες υποδομές που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανταλλαγή και την διαβίβαση, τη μεταφορά της ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο του κειμένου να μιλήσουμε και για τις τοπικές κοινότητες και το ρόλο τους σε σχέση με αυτές τις υποδομές. Σας ευχηστώ την προσοχή σε αυτό το σημείο, ε, ε, το σημείο ε, τις τοπικές κοινότητες. Ε, η, τα εμπορικά συμφέροντα θα επηρεάσουν τις ε, τοπικές κοινωνίες, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και την εκπαίδευση που κάνουμε σε αυτές τις κοινωνίες. Αν δεν υπάρχει συνένεση, αν δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, ε, μπορούμε να έχουμε προβλήματα με εγκληματικές οργανώσεις και να διεισδύσουν σε τέτοιες ε, τοπικές κοινότητες. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την ανάπτυξη ε, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην, ε, τις θέσεις απασχόλησης. Σας ευχαριστώ με αυτά ε, ακόμα μια φορά κύριε Μπούχνερ και όλους σας για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς τώρα θα λάβετε τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η εκθέση επιθυμεί να δώσει ακόμη περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ενέργειας και να αφαιρέσει εξουσίες από τα κράτη-μέλη. Θέλει να περάσουμε σε μια ευρωπαϊκή αγορά και διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές ε, βλέπουμε ότι δεν θέλετε πια να αγοράσετε φυσικό αέριο από τη Ρωσία το οποίο θα ικανοποιήσει σίγουρα την Αμερικανική κυβέρνηση στην ε, σταυροφορία που διεξάγει κατά αυτής της χώρας θα φέρετε με εισαγωγή το υγροποιημένο και πολύ ακάθαρτο ε, σχιστολιθικό φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ το οποίο θα έρχεται από τις, ε, με, με πλοία υψηλού κόστους. Δυστυχώς για εσάς οι χώρες με τις πιο ανταγωνιστικές αγορές είναι και εκείνες όπου οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλότερε. Η Γαλλία προσπαθεί να πάψει αυτή την, το, το ψευδή ανταγωνισμό, έχει τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Από την άλλη είναι σαφές ότι ορισμένα πυρηνικοί αντιδραστήρες όταν τους διαχειρίζεται μια δημόσια επιχείρηση ε, έχουν χαμηλότερη ε, αποδοτικότητα θα ήταν όμως πολύ επικίνδυνο να δώσουμε τη διαχείριση τέτοιων πυρηνικών αντιδραστήρων στον ιδιωτικό τομέα. Ξεχνάμε απόλυτα το πρόβλημα των οικονομιών κλίμακας. Αναφέρομαι εδώ στα φωτοβολταϊκά κέντρα η παραγωγή ενό συλλέκτη 10 ε, ε, τετραγωνικών μέτρων κοστίζει πολύ ψηλό. Πολύ οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση προς ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας είναι υψηλέ και δεν μπορούν να υλοποιηθούν εύλογα από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορεί να οδηγήσουν μάλιστα σε αύξηση κατά 5% των τιμών αυτών των ενεργειών. Οι καταναλωτές θα βρεθούν σε αδύναμη θέση ε, από τις ιδιωτικές εταιρείες και έτσι οι τιμές θα αυξάνονται αδιάκοπα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σίγητα, οι προτάσεις σας λοιπόν δεν έχουν καμία συνοχή. Θα οδηγήσουν σε πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα με λιγότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμε πηγές και ε, μείωση υποβάθμιση της δημόσιας ασφαλείας. Στούμε, Παρακαλώ εσείς Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να επισημάνω ότι είναι πολύ σπουδαία αυτή η γνωμοδότηση ως θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Έκανε πολύ καλό έργο συντάκτης της γνωμοδότησης και τον συγχαίρω και συμμερίζομαι για το θέμα των τροπολογιών που θα υποβληθούν από πλευράς ΛΑΝΕ. Κάποια στοιχεία της έκθεσης θέλω να τα εξετάσουμε για να εξειδικευθούν περισσότερο τα μέτρα που πιστεύω πρέπει να ενδυναμώσουμε. Αναφέρουμε ότι, στο ότι είναι σημαντικό να αναθεωρηθούν οι στόχοι της αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα, κράτη, μελη Πρέπει να κάνουμε βήματα, να πάμε πιο πέρα ε, όσον αφορά την φιλοσοφική προσέγγιση και τα σχέδιά μας ε, και ποσοτικά. Επίσης είναι σημαντικό να στο, ε, θεσπίσουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την ε, διασύνδεση μια τέτοια ενεργειακή ένωση χωρίς διασύνδεση που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά δεν θα είναι μια αυθεντική ενεργειακή ένωση και δεν μπορούμε για τον 21ο αιώνα να μιλάμε για μια τέτοια ένωση χωρίς την ενεργειακή ένωση και τη διασύνδεση αυτή και κάτι άλλο που συνδέεται άμεσα με τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την πολιτική εμπορικής προστασίας ώστε να υπάρξει διασυνοριακά ένας μηχανισμός που θα αφορά τα απαιτούμενα. Αν οι δικές μας ε, βιομηχανίες πρέπει να είναι ε, ανταγωνιστικές και πρέπει να είναι, πρέπει να είναι ανταγωνιστικές με μια προοπτική αηφόρου ανάπτυξης, με την προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες δίκαιους του παιχνιδιού που με αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιοι και να δούμε ότι εισάγονται προϊόντα που δεν υλοποιούν τις απαιτήσει που εμείς έχουμε θεσπίσει για τις επιχειρήσεις μας. Και τέλος, παρότι δεν είναι ένα θέμα οικονομικό και είναι θέμα αρχών, πιστεύω ότι στην γνωμοδότησή μας θα πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Ευχαριστώ. Äh, Σε ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τώρα τον λόγο. Ο κύριος Μάρτιν Βέστροπ, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλη την Επιτροπή για τη συζήτηση αυτή. Κυρίως ευχαριστώ για τη σύνταξη της γνωμοδότηση αυτής για τη σημαντική πρωτοβουλία. Η ενέργεια, η ενέργεια είναι μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, όπως συμφωνήθηκαν, συμφωνήθηκε από όλου πέρυσι και το εμπόριο στην ενέργεια είναι πολύ σημαντικό, ε, αν θέλουμε να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε ευγνώμονες που αποφασίσατε να συντάξετε μία γνωμοδότηση και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Ήτρε θα τη λάβει σοβαρά υπόψη να τα φτάσει μπροστά τη. Πολύ σύντομο θα είμαι. Θέλω να αναφέρω ένα-δύο σημεία ε, στο σχέδιο γνωμοδότηση που σχολίασαν και οι ευρωβουλευτές. Υποστηρίζουμε εν γέννη το σχέδιο που παρουσίασε ο εισηγητής. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε το πώς μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανανεώσιμης ενέργειας να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την εισαγόμενη ενέργεια. Αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε εξαρτώμενοι από αυτές τις εισαγωγές τα επερχόμενα χρόνια και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσουμε αυτή την αγορά ενέργειας, ούτως ώστε να, είμαστε, ε, να είναι σίγουροι, βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ενεργειακές συμφωνίες μέσω του εμπορίου, δηλαδή εμπορικές συμφωνίες για την ενέργεια και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη σας επί του θέματος αυτού, επί του σημείου αυτού. Το άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι του χρόνου θα εξετάσουμε μία... θα κάνουμε μία αναθεώρηση της απόφασης IGA, δηλαδή της διαθεσμικής ε, συμφωνίας, για την ενέργεια. Εν για να εξασφαλίσουμε ότι η ισχύουσα συμφωνία είναι απόλυτα συμβατή και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την απόφαση αυτή στο μέλλον μέσω της αναθεώρησης. Επίσης, θα ήθελα να πω για την επερχόμενη αναθεώρηση της, του καονισμού για το φυσικό αέριο, ότι θα εξετάσουμε τα θέματα που συνδέονται με τη διαφάνεια στις εμπορικές συμβάσεις και ε, τις κοινέ αγορές. Σας ευχαριστώ ακόμα μια στιγμή για το σχέδιο γνωμοδότησης. και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σας. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε κύριε Βέμπστρομ. Αναφερθήκατε στην, στο αναθεω... στην αναθεώρηση του κανονισμού για τη διαθεσμική συμφωνία. Αυτή η αναθεώρηση της συμφωνίας της διαθεσμικής ε, προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Θα μπορούσα να σας πω δύο λόγια, αλλά θα ήταν πρόωρο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα μαζί. Η Κομισιόν θα κάνει και μια πολύ ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, ούτως ή άλλως, και σε αυτή τη φάση δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη προς τα που θα κινηθούμε. Όπως είπα, όπως υπόθηκε και στην ανακοίνωση του Φεβρουαρίου για την ενέργεια, θα προσπαθήσουμε να έχουμε πριν συναφθούν αυτές οι συμφωνίες ως Κομισιόν πιο ισχυρό ρόλο. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα αυτή τη στιγμή να μας κοινοποιούν τις συμφωνίες που έχουν, θα τις εξετάσουμε. Αλλά όπως υπόθηκε και στην παρέμβασή σας, ε, το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε από την αρχή αυτές τις διαθεσμικές συμφωνίες. Θα τα εξολογήσουμε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να σας πούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι πολύ προωρό αυτό. Και τώρα κύριε Μπούχνερ, παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Φυσικά θα προσπαθήσω στο μέτρο του εφικτού να εντάξω τις προτάσεις σας και να βρούμε συνενετική θέση για αυτές. Προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία και τις νέες καλές ιδέες. Ευχαριστώ. Good. Πολύ καλά. Να επισημάνω κάτι, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 17η στις 12 το μεσημέρι. 17, 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στις 22 Σεπτεμβρίου. Πολύ καλά. Και έτσι περνάμε στο σημείο 10 τώρα την έκθεση για την αντιπροσωπεία στην Ιταλία, στη Γένοβα και Μιλάνο. Η αντιπροσωπεία υπό δύο προσεγγίσεις ε, έδρασε για τον, να δει τι γίνεται με τα λιμάνια στη Γένοβα και τα θέματα των λιμένων και δεύτερον στο πλαίσιο της έξπο της έκθεσης στο Μιλάνο να εξετάσει το θέμα της εμπορικής πολιτικής και των γεωργικών προϊόντων, αηφόρων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την ασφάλεια και την επισητιστική κάλυψη και να τα συζητήσει αυτά. Ο κύριος Κασπάρη, ο κύριος Φίσας, Ντάντι Μόσκα, η κυρία Μπεγκίν συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλες όλους που ενεργά συμμετείχαν και πιστεύω ότι ήταν μια καλή αποστολή αυτή η αντιπροσωπεία που σημαντικά θέματα εξέτασε στο λιμάνι της Γένοβας είχαμε επαφές με τις λιμενικές αρχές, ιδιαίτερα και με τις τελωνιακές αρχές, για να δούμε τι γίνεται με τα τελωνιακά θέματα και φυσικά και με τις αντίστοιχες, ε, ε αντίστοιχους εκπροσώπους βιομηχανιών και επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των προκλήσεων για τα θέματα φωτοεκφόρτωσης σε λιμάνια και να δούμε τι γίνεται με τις σχετικές διεργασίες και με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και στην ΕΞΠΟ με τα θέματα επισητιστικής ασφάλειας και τροφίμων και την κάλυψη των αναγκών μας επισητιστικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάναμε συζητήσεις, είχαμε επαφές και επισκεφθήκαμε και είδαμε για να ενημερωθούμε πώς ε, παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διεθνή έκθεση του Μιλάνου. Και στη συνέχεια και σε συζήτηση που είχαμε με εκπροσώπους του τύπου και πολίτες ανταλλάξαμε απόψεις, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις όλος ο τομέας αυτός ε, των θεμάτων πρόσβασης ε, στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα θέματα των προδιαγραφών για την ασφάλεια, ακόμα και τελωνιακή δασμοί γεωργικών προϊόντων μέσω των trade facilitations, των μέσων διευκόλυνσης ε, του εμπορίου και τις ποσοστώσεις και τα θέματα προστασίας αποτελούν και αυτά ένα ζήτημα που εξετάσαμε και υπό το πρίσμα της ε, Ιταλικής ε, αγροβιομηχανίας. Τα είδαμε αυτά και είχαμε και τη δυνατότητα τοπικά και περιφερειακά να συναντήσουμε εκπροσώπους, κυβερνητικούς εκπροσώπους και εκπροσώπους των περιφερειών και των τομέων και διεξαγάγαμε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Last Call Ευρώπη 2020 τελευταία κλίση, η αναγγελία για την Ευρώπη του 2020 και για την αηφορία ευθύνη των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο επίτευξης της Ευρώπης 2020 και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και είχαμε και χρόνο για τις ε, συζητήσεις και επαφές αυτές. Σημαντικό ήταν ότι σε αυτή την αντιπροσωπεία η συνεκτικότητα και η συνάφεια είναι κάτι που λάβαμε υπόψη από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βιομηχανίας και από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γεωργίας είχαμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε. Δεν είχαμε δηλαδή τρεις διαφορετικές αντιπροσωπείες, αλλά μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο παρουσιαστήκαμε. Αυτά από πλευράς μου εισαγωγικά. Την έκθεση την έχετε στα χέρια σας. Θα ρωτούσα από τα μέλη της αντιπροσωπείας υπάρχουν κάποιες συμπληρώσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Κύριε σας παρακαλώ και τον... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία, πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί με τη συνάδελφο την Τιτσιάνα Μπεγκίν ε, πήγαμε στο λιμάνι της Γένοβας, το επισκέψαμε. Μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά και οι λιμενικές αρχές καλά, καθώς και οι επιχειρηματίες. Και όπως λέγεται και στην έκθεση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξαναδούμε το πρόβλημα που υπάρχει με τα τελωνία. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία ε, ελέγχονται διαφορετικά από τελωνία σε τελωνία ανάλογα με το που εισάγονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια ας πούμε ιταλικά προϊόντα, κάποια τυριά ας πούμε ιταλικά, τα οποία εισάγονται από τις Φιλιππίνες ε, εισάγονται στις Ηνωμένε Πολιτείε χωρίς επαρκή έλεγχο, κυρίως του, της ονομασίας προέλευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το μελετήσουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Επίσης, μαζί με την κυρία Μπεγκίν θέλουμε να παρουσιάσουμε μία πρωτοβουλία, να κάνουμε μία ακρόαση δηλαδή, για τα λιμάνια στην Μεσόγειο και την διασύνδεση, το πώς συνδέονται μεταξύ τους και τον, τα βόρεια λιμάνια αλλά και πώς συνδέονται ας πούμε με τα λιμάνια της Αφρικής και της ε, Ασίας. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών και είναι μια πρωτοβουλία που θα την υποβάλουμε πολύ σύντομα. Frau σε ευχαριστούμε κυρία Ντεσαρνές παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τους βουλευτές που μετέβησαν στο λιμάνι της Γένοβας και να μου πούν πώς είναι τα πράγματα επιτόπου όσον αφορά τους ελέγχους. Πράγματι ελέγχονται τα τρόφιμα, ελέγχονται οι γεωγραφικές ενδείξεις. Αν ναι, ποιο ποσοστό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που υπάρχουν ε, για να επιτραπεί η είσοδο του ε, στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Ευχαριστώ πολύ. Α, θα ήθελα αυτέ τι εξηγήσει. Perdón. Sí es cierto que mm, hay veces que no se... δεν γίνονται έλεγχοι με τον καταλληλότερο τρόπο. Αυτό είναι σίγουρο. Εξαρτάται από το είδος του προϊόντος. Μερικέ φορέ γίνεται ένα τελώ αφαίρετο και τυχαίο έλεγχο. Φυσικά δεν, γίνεται δυνατό, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε έλεγχο σε όλα τα προϊόντα. Επομένω, τυχαία διαλέγουν κάποια προϊόντα και τα ελέγχουν. Και δυστυχώ, κάποια προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να μπουν στην Ευρώπη μπαίνουν. Επίσης, επιμένουμε πάρα πολύ στον έλεγχο τη ονομασία προέλευση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος. Αυτός, αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο το λιμάνι της Γένοβας, αφορά όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Έχουμε δεδομένα από προϊόντα, δεν θυμάμαι, ας πούμε, ιταλικά τυριά, δεν θυμάμαι ποιο ιταλικό τυρί, που μας είπαν Μας έδειξαν και κάποια έγγραφα για αυτά τα, προϊόντα. Ότι μπαίνουν σε κάποια λιμάνια ευρωπαϊκά χωρίς να ελέγχεται η ονομασία προέλευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και η προλαλήσασα. Και θα πρέπει στο μέλλον να, το, να μας απασχολήσει πραγματικά σοβαρά το θέμα του ελέγχου και να εμποδίσουμε αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι προϊόντα απομιμήσεις των ευρωπαϊκών προϊόντων, να ξαναμπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά ε, μέσω των λιμανιών μας, λόγω αυτού του προβλήματος των ελέγχων. Um, Αυτό το θέμα που αναφέρατε είναι πολύ καλό. Το θέμα των τελωνιακών <clears throat> ελέγχων και διαδικασιών Αποκινούμε την Επιτροπή Μεταφορών νομίζω μπορούμε να δώσουμε συνέχεια με δική μας πρωτοβουλία και για το θέμα της κυρίας Δεσαρνές στην έκθεση αναφέρονται κάποια στοιχεία ότι 37% των απομιμήσεων προέρχονται από μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποια είναι αλλά και άλλα στοιχεία θα υπάρχουν ώστε να προχωρήσουμε πολύ καλά Υπάρχουν ε, άλλες επερωτήσεις ή άλλα σχόλια για την αντιπροσωπεία μας που πήγε στη Γένοβα και στο Μιλάνο. Παρακαλώ. Όχι, δεν υπάρχουν. Ώστε θα διακόψουμε τώρα τη συνεδρίες για έξι λεπτά ακριβώς. Θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Good. Mm, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι. Α συνεχίσουμε τη συνεδρίαση και περνάμε στο σημείο 11 την ψηφοφορία που αφορά το τριμερή διάλογο για τα μέταλλα από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού Αφορά επίσης και τη σύνθεση της αντιπροσωπείας. Έχουμε ήδη αναβάλει τη ψηφοφορία και στο μεταξύ ο πρόεδρος, η πρόεδρος το μελέτησε και συνέστησε να ακολουθήσουμε το, η παραδοσιακή οδό και να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο. Θα έχετε λάβει τον καταλόγο ψηφοφορίας, τη λίστα ψηφοφορίας όσον αφορά την αρχή του τριμερούς διαλόγου αλλά και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως ξέρετε στο άρθρο 73 το ζήτημα ρυθμίζεται στο άρθρο 73 όπως το ζήτημα της σύνθεσης των στόχων της ε, παραπομπής στην Επιτροπή και μετά η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής ε, που πρέπει να αποφασίσει την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων και τη σύσταση αυτής της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων. Αυτά είχα να πω εισαγωγικά. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ich habe hier 39 Stimmkarten und jetzt haben auch 39 Kollegen. 39. Και βλέπω ότι ψήφισαν 39 συναδέλφοι, οπότε όλα λειτουργούν. Έχουμε ολοκληρώσει την ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Μια χαρά. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για την έναρξη του τριμερούς διαλόγου και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Άρχεται η ψηφοφορία. Und die Abstimmung ist Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρα. και 15 εποχές. Οπότε θα ακολουθήσουμε. Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 12. την ε, έκθεση που αφορά τις ε, ανταλλαγές ε, του Μπαλή, τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 31 1 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές για άλλη μια φορά τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβεβαστική 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπ... εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβεστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δευε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεβεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist Πέρας ψηφοφορίας. Πρέπει να πω ότι κάποιοι δεν ήταν πολύ σαφείς πριν. Έγκρινεται. Σε κάθε περίπτωση τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 Ah, Ξέχασα, λέει ο Πρόεδρο, την 13. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 13 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου άρχεται ψηφοφορία Abstimmung ist ψηφοφορίας 29 υπέρ 4 κατά 6 αποχές συγχαρητήρια Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 13 σχετικό το ζήτημα με το 12. Εάν δώσουμε τη συμφωνία μας εδώ για αυτή τη διευκόλυνση του εμπορίου, ε, για να δώσουμε τη διευκόλυνσή μας, είναι μία ψηφοφορία μόνο για το σύνολο, άρχεται η ψηφοφορία. Und Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Ευχαριστούμε για την ταχύτητα της ψηφοφορίας. Έχουμε λοιπόν, είμαστε ένα τέταρτο μπροστά σε σχέση με το επόμενο σημείο, αλλά σας παρακαλώ μην φύγετε διότι 10 και μισή θα ξεκινήσουμε με την ακρόασή μας, η οποία